με τις θέσεις αυτές που είπατε. Δεν νομίζω να υπάρξει κανένα είδους πρόβλημα. Όσον αφορά την επιλογή διορισμό των υποψηφίων. Ευχαριστώ πολύ και τώρα στην εμέρεση διάταξη έχουμε την κοινή συζήτηση για το θέμα της μπανάνας. Έχουμε καταρχάς μια σύσταση κυρίας Βαρτζάνη για το εμπόριο και μετά έκθεση για την κατάργηση του κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τους δασμούς για τις μπανάνες. Και επιπλέον έχουμε προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τις συμφωνίες για το εμπόριο μπανάνες. Η κυρία Παλτσάνη ως εισηγήτρια θα λάβει το λόγο για τις δύο εκθέσεις και εκ μέρους της Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου. Θα τοποθετηθεί και για τις προφορικές ερωτήσεις και θα έχει χρόνο ομιλία τόσο στην αρχή σου και στο τέλο τη συζήτηση. Έχετε καταρχάς το λόγο για έξι λεπτά κυρία Παλτζάνη. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το Κοινοβούλιο καλύτερα να τοποθετηθεί επί δύο συμφωνιών που υπεγράφησαν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με 11 χώρες της Λατινικής Αμερικής και που έρχονται για να δέσουν τέλος σε μια μακροχρόνια υπόθεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ΠΟΕ ε, σκέφτηκε δίωξη για της ευρωπαϊκές Ένωσης στα πλαίσια του ΠΟΕ. Το θέμα είναι πάρα πολύ λεπτό γιατί οι διαφορές ε, αφορούσαν την αρχή τη μη εισαγωγή διακρίσεων στις ε, διεθνεί Εμπορικέ σχέσεις ε, που αντίθετα η Ευρώπη θα είχε παραβιάσει ε, κατά την ε, οργάνωση εισαγωγή μπανανών στο εσωτερικό της Ένωσης. Αυτό οφείλεται σε ένα διτό σύστημα που εφαρμόστηκε εναντί των χωρών ΑΚΕ, εναντί άλλων χωρών ένα σύστημα το οποίο επέτρεπε στις χώρες ε, αυτές ε, να εισάγουν ε, αυτά τα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αδασμολόγητα σε αντίθεση με άλλες χώρες που έπρεπε να καταβάλουν δασμούς για 176 ευρώ ανά τόνο. Με αυτή τη συμφωνία λοιπόν ε, έρχεται νέα ισορροπία στην κατάσταση και καταρχήν διατηρείται το δικαίωμα των χωρών και που είναι ε, χώρες αναπτυσσόμενες σε λεπτή κατάσταση ανάπτυξης να εισάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα προϊόντα τους δίχως να καταβάλουν εισαγωγικού δεσμούς. Παράλληλα, οι υπόλοιπε χώρες που υπέγραψαν τις συμφωνίες ε, θα μπορούν να εξάγουν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπανάνες πληρώνοντας πάντα δασμούς αλλά που θα μειωθούν ε, σε μια χρονική περίοδο από το 2011 ως το 2017 δηλαδή προοδευτικά ε, από τα 176 ευρώ τον τόνο στα 114 ευρώ τον τόνο. Αλλά το πιο σημαντικό αυτών των συμφανιών είναι πέρα από το ότι τελικά ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρεί τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στα πλαίσια του ΠΟΕ κατά κάποιο τρόπο αποκαθιστά και μια θεσμική αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πέραν αυτού ε, οι αναπτυσσόμενες χώρες ΑΚΕ λαμβάνουν ιδιαίτερη προσοχή γιατί προβλέπονται μαζί με τις συμφωνίες και νέα μέσα χρηματοοικονομικής στήριξης υπέρ τους. Αυτά τα μέτρα χρηματοοικονομικής στήριξης θα επιτρέψουν στις χώρες αυτές να επενδύσουν για να διαφοροποιήσουν την παραγωγή τους Επομένω, επομένως για να ενισχύσουν και την οικονομία τους ως ευκταίο. Αυτά τα μέτρα έχουν ε, ένα ε, βάρος ε, περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ και πλευρέποντας το 2013. Αυτές οι συμφωνίες λοιπόν θεωρώ ότι είναι θετικές όχι μόνο γιατί ε, θέτουν τέλος σε διαφορές ε, που θα βάρυναν ε, οικονομικά την Ένωση και με κυρώσει, αλλά και θα έθεγαν τη θεσμική τη αξιοπιστία, αλλά και γιατί επιτρέπουν την εξέβρεση μια ισορροπημένη λύση και έναντι των χωρών ΑΚΕ και έναντι των Ευρωπαίων παραγωγών στι ε, πλέον απομακρυσμένε περιοχέ που σίγουρα δεν μπορούν να εγκαταλειφθούν σε έναν αφέμητο ανταγωνισμό, σε έναν αγριό ανταγωνισμό και γι' αυτό το Κοινοβούλιο προτείνω να δώσει την έγκρισή του σε αυτές τις συμφωνίες τα όμως από την Κομισιόν και το Συμβουλίο να δεσμευτούν για να ε, προβούν σε μία ε, αξιολόγηση αντικτύπου αυτών των συμφωνιών ε, ως το 2020 σε έναν ευρύ ερίζοντα τις συνέπειες λοιπόν που θα υπάρχουν και στις χώρες εκεί αλλά και στους ευρωπαϊκούς παραγωγούς όταν η οικονομία ε, κάποιων περιφερειών, όπω των πλέον μικρών περιοχών, συνδέεται με την παραγωγή αυτοπροϊόντο, αλλά επίση να δεσμευτούν πριν να ολοκληρωθούν ε, τα, πριν να ολοκληρωθεί η λειτουργία του ε, μέσου, του δικού μηχανισμού που χρησιμοποιείται για τι χώρε ΑΚΕ, να δεσμευτούν η Κομισιόν και το Συμβούλιο να προβούν σε μια αξιολόγηση τη λειτουργία των μέτρων αυτών χρηματοοικονομική στήριξη 18 ε, μήνε πριν από ε, τη λήξη του προγράμματο, έτσι ώστε να μπορούν ενδεχομένως να παρέμβουν με ένα άλλο μηχανισμό στήριξης ε, των χωρών αυτών γιατί ε, ακριβώς ε, δεν πρέπει να, ληφθούν, να μόνες και πρέπει να υποστηριχθούν για να μειώσουν τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες που θα προκύψουν από αυτές τις συμφωνίες με μια διόρθωση των τιμών της ανταγωνιστικότητας των που προέρχονται από τις άλλες χώρες. Ε, έτσι λοιπόν πιστεύω ότι είναι μια συμφωνία που αυτή τη στιγμή επιτρέπει να βρούμε μία διέξοδο σεβόμενη και αυτές τις πιο αδύναμες χώρες. Και επαναλαμβάνω, αυτή ήταν η κύρια ανησυχία που κατά τη διάρκεια της μακράς συζήτηση που είχαμε στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ε, πάντοτε ε, είχαμε κατά νου και εύχομαι να μπορέσει να ε, τύχει ισχυρή στήριξη και αναφέρομαι κυρίως ε, στις δεσμεύσεις που ζητάμε εμείς να αναλάβουν η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Πρέπει η Κομισιόν και το Συμβούλιο να υποπτεύουν αυτή τη συμφωνία και να προβούν και σε ενδεχόμενη ενίσχυση για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπαλτζάνη. Τώρα κυρία Ζωρή εκ του Συμβούλιο και πάλι. Παρακαλώ. Γερ. Στα Ιταλικά λέει ευχαριστώ. Για τώρα, ε, τον κύριο Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ και κυρία Συγγετρία Μπαλτσάνη, σα ευχαριστώ τόσο πολύ διότι μου δώσατε την ευκαιρία. Γιατί μου δώσατε την ευκαιρία να παρέμβω σε ένα σημαντικό θέμα τόσο από τη σκοπιά του διεθνούς εμπορίου όσο και από τη σκοπιά της αλληλεγγύης και της ανάπτυξης. Ε, ελπίζω να μπορέσω να απαντήσω στις ερωτήσεις ε, κ. Μορέιρα αλλά και τις, ε, στις ανησυχίες που αναφέρθηκαν από την κυρία Μπαλσάνη. Και αν επιτρέπετε θα συνεχίσω στα ογκρικά. Και το Συμβούλιο έχει πλήρη επίγνωση του ότι ε, πρόκειται για θέμα μεγάλης σημασίας οικονομικής και κοινωνικής εκεί όπου παράγεται η μπανάνα. Αυτό έχει να κάνει με την επιβίωση των παραγωγών, οπότε και γι' αυτό θα πρέπει να κάτσουμε και να κάνουμε μια αξιολόγηση αυτών των συνοδευτικών μέτρων και αυτό θα πρέπει να γίνει 18 μήνες πριν σταματήσει να τρέχει η εκπνεύση διάρκεια του προγράμματος και κυρίες και κύριοι ξέρουμε ότι ότι η αξιολόγηση αυτή αλλά και η περαιτέρω προτάσεις είναι αρμοδιότης της Κομισιόν και όχι του Συμβουλίου. πάντως ελπίζουμε ότι ο αρμόδιο συνάδελφο πρόκειται να τα φροντίσει αυτά και ο πρώτο επίτροπο. Οπότε και ε, λαμβάνω υπόψη αυτό που είπα στην προφορική σα την ερώτηση για τις αξιολογήσεις και για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα συνοδευτικά μέτρα θα πρέπει να λάβουν υπόψη τι γίνεται με τις καλυπτόμενες χώρες τι επιλέξιμε τέλο πάντων, τόσο ώστε θα πρέπει να επιλύσουν τα θέματα που ακόμα εκκρεμούν, ώστε να μην καθυστερήσει η λήψη αυτό το μέτρο Τώρα, όσον αφορά την κατανομή των σχετικών πόρων για τα συνοδευτικά μέτρα το Συμβούλιο ήταν υπέρ του σχεδίου εικονισμού όσον αφορά αυτά τα συνοδευτικά μέτρα. Και η πρώτη ανάγνωση, ο δε ε, κανονισμός αυτός ορίζει κατά τα κριτήρια, τους δείκτες, τις μεταβλητές, τόσο ώστε να ληφθεί υπόψη ο όγκος της συμπορικής ροής αυτών των προϊόντων την υπόψη σημασία για τις χώρες και αλλά και το νοτισιακό επίπεδο της ε, κάθε φορά εξεταζομένης χώρας. Στις 24 Σεπτεμβρίου πέρυσι είπαμε ότι 6% των μέτρων των, των πόρων αυτών πρόκειται να πάει στις περιοχές απότερες περιφέρειας της ε, Ένωσης και όσον αφορά για τις συμφωνίες ελευθερών εμπορίου με την Κολομβία, το Περού και τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής έγιναν κάποιες επαφές για την μπανάνα με την ε, Κομισιόν στα πλαίσια των συμφωνιών πλαίσιο αλλά ακόμα δεν υπάρχει επίσημη θέση, δεν μπορώ να σου πω τίποτα με την κοινότητα των Άνδρων επίσης έχουμε επαφές και διπλωματεύσεις ώστε να υπάρχει κάποιο είδους διαπεριφερειακή συμφωνία. Όμω διακόπησαν οι διαπραγματεύσει τον Ιούνιο του 2008 γιατί δεν συμφωνήσαμε για τα εμπορικά θέματα. Οπότε μετά όμω, τον Ιανουάριο του 2009 συνεχίστηκαν οι διαπραγματεύσει με Κολομβία και Περού. Τόσο να υπάρξει μια πολυμερή εμπορική συμφωνία ελευθέρω εμπορίου. Το Εκουαδόρ απεσύρθε τον Ιούλιο του 2009 διαπραγματεύσει με Περού και Κολομβία πάντω συνεχίστηκαν εκ τότε και ολοκληρώθηκαν και οι συνομιλίε που έκανε η Κομισιόν με αυτέ τι δύο χώρε την 1η Τρίτου του 2010. Και έχουμε άλλε χώρε τη Κοινοδοσυνάδεων που είναι το Εκουαδόρ και που μπορεί όποτε θέλει να προσυπογράψει τη σχετική συμφωνία. Και έτσι έχει δηλωθεί επίσημα τη χώρα αυτή ότι προτίθενται να συνεχίσουν τι επαφέ και εμεί θεωρούμε ότι είναι αυτό πάρα πολύ θετικό. Και αν ξεκινήσουν αυτέ οι επαφέ με το Εκουαδόρ, τότε θα πάμε σε μεγάλο όγκο συναλλαγών, θα φτάσουμε στους στόχους που έχουμε τάξει για τις εμπορικές μας σχέσεις με αυτές τις χώρες, οπότε παρακαλώ αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, δώστε το πράσινο φως για αυτές τις συμφωνίες και παρακαλώ επίσης δώστε το πράσινο φως ούτως ώστε να ανασταλεί η σχέση του κανονισμού που αφορά τους δασμούς της μπανάνας και εμείς υπολογίζουμε στην βοήθεια και συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιώρη Εκ μέρους Επιτροπής. Ο αρμόδιο επίτροπος, κύριος Τσόλος, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρία Παλτσάνη, κυρίες και κύριοι. Με ικανοποίηση καταρχάς διαπιστώνω ότι οι κύριες Πτυχε και οι κατευθύνσεις τον των, των θέσεων τη Επιτροπή για την Μπανάνα την χάνουν τη συμφωνία της εισηγητρίας. Η κυρία Παλτσάρη με πολύ εύστοχο τρόπο παρουσίασε και το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν αυτέ οι διαπραγματεύσει και συνήφθη η συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρί επιφύλαξη, υποστηρίζει το σχέδιο συστάσεων τη ε, κυρία Συγητρία, καθώ και το σχέδιο εκθέσεω για το ίδιο θέμα. Οι συμφωνίε τη Γενέβη του 2009 για την παρανένα ασφαλώ πολύ σημαντικέ, όπω πολύ εύστοχα επεσήμανε και εξήγησε η κυρία Βαλτσάνη, και θα ήθελα επίση να υπογραμμίσω ότι αυτέ οι συμφωνίε θα φέρουν πλέον ε, την ειρήνη σε αυτό το ακαθόδε ζήτημα και θα διευκολύνουν τη διαδικασία της ΔΟΧΑ, ορίζοντας στο ε, προϋποθέσεις για την θέσπιση μιας αγοράς ευρωπαϊκής της ε, μπανάνας σταθερής και προβλέψιμης για τα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα τώρα να επανέλθω σε κάποια από τα σημαντικότερα ζητήματα που θίγονται από την εισηγήτρια και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προφορική ή τις γραπτές ερωτήσεις καθώς και στην πρόταση ψηφίσματος που συμπεριληφθεί σε αυτές τις προτάσεις όσον αφορά την υποστήριξη, τη στήριξη μάλλον στους παραγωγούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελώ γνώση του κοινωνικο-οικονομικού ρόλου και ρόλου για το τομέα τη παραγωγής μπανάνας, ιδιαίτερα στι άκρο ε, απομακρυσμένε περιοχέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως την ε, ζωτική σημασία για την επιβίωση αυτών των περιοχών ε, ε, το, το ρόλο ζωτική μπορεί που δραματίσει αυτό ο τομέα. Άλλωστε, έχουμε υποβάλει στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο του 2010 ανακοίνωση στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξηγεί τη σημασία και τι συνέπειε των συμφωνιών τη Γενέβη και το γεγονό ότι ήδη στη μεταρρύθμιση του 2006 το καθεστώτο που εφαρμόζεται στην Πανάνα έχει συμπεριληφθεί αυτό το νέο πλέγμα. Έτσι ώστε να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαδικασία της ε, ενισχυμένης απελευθέρωσης ε, της αυξημένης μονοπλευθέρωσης έχουμε ιδιαίτερα ε, λάβει υπόψη την ανάλυση επιπτώσεων, δηλαδή την ε, σημαντικότερη από, ό,τι τελικά συνήφθη, συμφωνήθηκε δηλαδή μείωση των τιμολογίων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαγρυπνά ώστε να προλαμβάνει δυσμενείς ενδεχομένως συνέπειες αυτών των συμφωνιών στις αγορές και αν χρειάζεται να λαμβάνει τα μέτρα ώστε να ε, μετριάσει αυτές τις δυσμενείς επιπτώσεις. Όσον αφορά την ενίσχυση της θέσεως των παραγωγών μπανάνας στην αλυσίδα της παραγωγής. Θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν πρόκειται για ένα ζήτημα που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα το τομέα της μπανάνας, αλλά έχει να κάνει με όλο τον τομέα το γεωργικό ε, της παραγωγής των τροφίμων, η θέση δηλαδή του παραγωγού στην αλυσίδα και ε, πόσο λόγο θα έχει ως προς την προσθέμενη αξία τη παραγωγή του στην ε, τροφική αλυσίδα είναι κάτι που αφορά ολόκληρο τον τομέα και στη μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική Πολιτική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις προσοχές της προτάσεις θα καταθέσει λύσει για την ενίσχυση του ρόλου των οργανώσεων παραγωγών σε αυτή την αλυσίδα και Τη της του τους ισχύω. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει μια υψηλού επιπέδου επιτροπή για την ε, αλυσίδα παραγωγής ε, γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ε, όπου συμμετέχουν πολλοί επίτροποι, και όχι μόνο ο Επίτροπος Αρμόδιο για τα γεωργικά θέματα που έχει περιορισμένες εξουσίε, αλλά και άλλοι τρει οι οποίοι καθοδηγούν τις εργασίε σε αυτή την ομάδα υψηλού επίπεδου. Ε, με προτάσεις ε, τις οποίες τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους επόμενους μήνες και έτη θα προωθήσει έτσι ώστε να δώσει απαντήσεις στο ζήτημα της διαφάνειας της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων. Και στο πλαίσιο αυτό ο παραγωγός πανάνας θα έχει τη θέση του, τη θέση που το αρμόζει στην αλυσίδα παραγωγή τροφίμων. Όσον αφορά τώρα την κατανομή των χρηματοπιστωτικών πόρων για τα συνοδευτικά μέτρα στο ζήτημα τη μπανάνα, στον τομέα τη μπανάνα, και τις χώρες της ΑΚΕ. Όπως γνωρίζετε το σχέδιο κανονισμού το οποίο προσδιορίζει αυτό που ονομάζεται BAM, δηλαδή τα στοδευτικά μέτρα, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 21 Οκτωβρίου. Προβλέπει αυτό το σχέδιο ε, λύσεις για την κατανομή αυτών των πόρων και κριτήρια συγκεκριμένα όπως τα ζητάτε. Ήδη περιλαμβάνονται στον κανονισμό αυτών. Εν προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάστηκε σε στενή συνεργασία και κατά τρόπο επικοδομητικό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να ετοιμάσει αυτά τα μέτρα και εξευρέθη μια ικανοποιητική συμβαστική λύση επί τη ουσία για πολλά από αυτά τα θέματα. Και το σχέδιο κανονισμού, το οποίο ιδιαίτερα ε, στοχεύει τα κράτη, και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προσδιορίζεται ταυτόχρονα και τα κριτήρια κατανομή για τα διάφορα δικαιούχα κράτη, ταυτόχρονα όμως και προσδιορίζοντας, όπως ε, αναφέρατε και εσείς, ότι πρόκειται να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης των αγορών στις χώρες αυτές 18 μήνες πριν από την εκπνοή του προγράμματος. Με την αξιολόγηση αυτή θα μπορέσουμε να κρίνουμε εάν έχουν υλοποιηθεί σωστά οι διαδικασίες προσαρμογής ή αν ενδεχομένως χρειάζονται άλλα μέτρα. Όσο τώρα αφορά την ανάλυση επιπτώσεων ως προς τις ε, συνέπειες αυτών των συμφωνιών σε και άκρως απομακρυσμένες περιοχές, και αξιοπροπισμένε περιοχέ τη Ευρώπη. Ήθελα να πω ότι βεβαίω αυτή η ανάλυση είναι πάρα πολύ απαραίτητη, αλλά α είμαστε και ρεαλιστέ προ το πεδίο που μπορεί να καλύψει μια τέτοια έρευνα, γιατί έχουμε να κάνουμε με πολλές χώρες στον κόσμο. Πολλές χώρες παραγωγού μπανάνας, πολλές χώρες για τις οποίες η μπανάνα είναι ε, βασική τροφή. Και άρα θα πρόκειται για μια μελέτη περίπλοκη και μια μελέτη της οποίας ε, η συναγωγή αποτελεσμάτων θα αποδειχθεί αρκετά επίπονη. Αλλά βεβαίω πιστεύουμε ότι μια μελέτη μπορεί να είναι χρήσιμη και μπορεί να στηριχθεί και σε μελέτε ε, και δεδομένα μελετών που έχει τη θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε εσωτερικέ είτε εξωτερικέ μελέτε. Και όπω είπα και νωρίτερα, θα προβούμε σε μια ανάλυση των συνεπειών των συνοδευτικών αυτών μέτρων για τα κράτη και 18 μήνε πριν από την εκπνοή του προγράμματο. Επίση, σε σχέση με την ε, ερώτηση σχετική με τη σύναψη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με ορισμένε χώρε τη Λατινική Αμερική και ειδικότερα του Εκουαδόρ. Ασφαλώ θα γνωρίζετε ότι η κατάσταση σχετική με τι εμπορικέ συμφωνίε με την Κολομβία, το Περού και τα κράτη τη Κεντρική Αμερική ολοκληρώθηκαν σε τεχνικό επίπεδο κατά τρόπο ε, ικανοποιητικό. Η συμφωνία με την ε, Κολομβία και το Περού είναι ανοιχτέ, μάλλον η συμφωνία είναι ανοιχτή και προ άλλα κράτη τη ε, συμφωνία των Άνδεων. Άρα Μπορεί και το Εκουαδόρ να προσχωρήσει και άλλωστε έχει ζητήσει το Εκουαδόρ να επανέλθει στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων προκειμένου να συζητήσει την ε, συμφωνία αυτή και η κυβέρνηση και οι αρχέ του Εκουαδόρ αυτή τη στιγμή εξετάζουν τι προποθέσει και του όρου ανάληψη των διαπραγματεύσεων και γενικά την πορεία που θέλουν να ακολουθήσουν. Αυτέ είναι οι ολίγε παρατηρήσει που είχα να κάνω σε σχέση με την έκθεσή σα, σε σχέση με τι ερωτήσει που υποβάλλατε. Ξέρω ότι μακρηγόρησα, αλλά ήθελα να δώσω στο δυνατόν πιο πλήρε απαντήσεις στην ερώτηση στο βαθμό που μου το επιτρέπει οι πληροφορίες μου. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ο εισηγητή τώρα εκ μέρου Επιτροπής ε, Αναπτύξεως, ο κύριο Γκέρνς για τρία λεπτά. Πρόεδρε, μεταξύ των ορίων του των αρχών του διεθνού δικαίου υπάρχει και η αρχή τη μη εισαγωγή διάκριση. Ε, θεωρητικά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, αλλά στην πράξη είναι διαφορετικά πράγματα. Οι ΑΚΕ ε, δεν καταβάλουν ε, εισαγωγικού δασμού για την εισαγωγή των προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και υπάρχουν συμφωνίε και δεν αλλάζει τίποτα. Όμω η μία ΑΚΕ πλήρωναν 176 ευρώ το τόνο τώρα και τώρα θα καταβάλουν δασμού μέχρι 141 ευρώ. Ε, δηλαδή ε, αλλάζει και η κατάσταση του ανταγωνισμού με τις μειώσεις αυτές. Ε, οι χώρες εκει ήταν πιο προστατευμένες τώρα, ενώ θα είναι λιγότερο στο μέλλον. Η Κομισιόν διαπραγματεύτηκε αυτή τη συμφωνία εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. στο θέμα είναι να ξέρω εγώ ω εισηγητή για τη γνωμοδότηση αν η Κομισιόν θα μπορούσε να πράξει διαφορετικά. Η απάντηση είναι σαφή, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, γιατί αν είχε κάνει διαφορετικά, αν είχε αρνηθεί να μπει σε αυτέ τι διαπραγματεύσει, θα είχε ρυθμιστεί το ζήτημα ε, στο όργανο επίλυση διαφορών του ΠΟΕ. Και τα αποτελέσματα εκεί φυσικά θα ήταν διαφορετικά από αυτά που αποκτήθηκαν ε, κατόπιν των διαπραγματεύσεων ε, της οποίες ε, συζητούμε. Δηλαδή τώρα ζούμε σαν έναν ιδανικό κόσμο, όχι εγώ είμαι εισηγητής για γνωμοδότηση, αλλά ε, είμαι και επί της ουσίας εισηγητής για μια έκθεση ε, για τον πόρο και έχω κάποια σχόλια να κάνω. Καταρχήν, ο προπολογισμό για τον τομέα της μπανάνας έχει αυξηθεί, το επενθύμησε και ο Επίτροπος ε, και έτσι απαντούμε και στην ερώτηση της κυρίας Σέντησες που ενισχύει πάρα πολύ για την κατάσταση που δημιουργείται για τους ε, παραγωγούς ε, μπανάνας από τις πλέον απομακρυσμένες περιφέρειες της ε, Ευρώπης. Ε, κύριε κυρία και εγώ είχαμε μια ακόμα ανησυχία ε, στην Επιτροπή Ανάπτυξη ότι με τα 114 ευρώ δεν τελειώνει εκεί η μείωση γιατί η Κομισιόν διαπραγματεύεται και άλλες συμφωνίες που πηγαίνουν πέρα από αυτά τα 114 ευρώ. Μιλάμε μάλιστα για 75 ευρώ. Έτσι λοιπόν ε, η μη διάκριση θα πρέπει να ακολουθήσει και αυτή την πτωτική πορεία. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό τρίτον σε ό,τι αφορά τα συνοδευτικά μέτρα για την μπανάνα και αύριο το πρωί θα μιλήσω πιο λεπτομερώς. Ε, νομίζω ότι το Κοινοβούλιο κατάφερε και ευχαριστώ τον Επίτροπο που αναφέρθηκε σε αυτό να εισαγάγει κάποιες καινοτομίες. Ε, αναφέρομαι συγκεκριμένα στην ε, μελέτη αντικτύπου 18 μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας του προγράμματος. Αυτό θα μας επιτρέψει να πάμε λίγο παραπέρα από το 2013 γιατί πιστεύω ότι το 2013 δεν θα έχει ολοκληρωθεί το πρόβλημα με τις τις μπανάνες. Ευχαριστώ και τώρα έχουμε τους ομιλητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Πρώτη εκ μέρους της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Δημοκρατών η κυρία Αντρική Ένε. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να επιθυμήσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο να δώσει το πράσινο φω στη σταθερή σημαντική συμφωνία, διότι θεωρούμε ότι έτσι πρόκειται να, να διευκολυθούν οι διαπραγματεύσει τη Ντόχα και επίση έτσι θα δοθεί νέα όθεση διμερεί επαφέ με τι χώρε Μερκοσούρ όσον αφορά την Συμφωνία Ελευθερού Εμπορίου και επίση θέλουμε να καλωσορίσουμε αυτή τη γενική τάση τη απελευθέρωση απορρίθμιση του εμπορίου Μπανάνα και επίση τη συμφωνία στα πλαίσια του ΠΟΕ αλλά και τι άλλε διμερεί συμφωνίε με τι χώρε των Άνδρων και τη Κεντρική Αμερική. και ίσω κάποια μέρα ακολουθήσει και ο Μερκοσούρ και τώρα έχουμε αυτό το ψήφισμα το οποίο είναι πάρα πολύ αξιόλογο, μπράβο στον εισηγητή και επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι λύθησαν υπόψη τα συμφέροντα των εταίρων μα από τι χώρε αλλά αλλά για των τοπικών παραγωγών μπανάνα. Ε, Εμεί έχουμε τη στρέπη επίθεση ότι όσο προχωράει η απορρίθμιση του πολύ μπανάνα θα πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι έτσι δεν θα αφανίζουν ολόκληροι τομεί, ολόκληρε βιομηχανίε που έχουν παραδοσιακά παίξει σημαντικό ρόλο στην κοινωνία και την οικονομία διαφόρων περιοχών όπως τη Γουαδελούπη, τη Μαρτινίκα, τα Κανάρια, την Μαδέρα, τις Αζόρες και αλλού. Επίσης τελικά συμφωνούμε ότι πρόκειται όλα αυτά να τα λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα αναλάβει τα απαραίτητα τόσο ώστε να μπορέσει να εγκρίνει αυτό το, το πακέτο μέτρων στήριξης των τοπικών παραγών. Και επίσης να λάβει τα απαραίτητα μέτρα στα πλαίσια του ΠΟΣΕ ούτως ώστε να προχωρήσει η απορρίθμιση. Και οι δικοί μα παρόκειται να μείνουν μέσα στην αγορά, να συνεχίσουν τι προδιαστικές δραστηριότητε. Είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη ευκαιρία που θα προκύψει κατά τι συζητήσει για τι μελλοντικέ δημοσιονομικέ προοπτικέ. Σα ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Εκ μέρου τη Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να μιλήσει τώρα ο κύριο Τιγολιά. Δεν τον βλέπω όμως στο ημικύκλιο και γι' αυτό δίνω το λόγο στον επόμενο ομιλητή από τους Σοσιαλδημοκράτες, τον κύριο Αρσένη παρακαλώ. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά κύριε Αρσένη. Η έννοια των ε, Banana Republics, των μπανανιών, είναι γνωστή σε όλους μας. Είναι όλες αυτές οι χώρες όπου οι μεγάλες εταιρείες παραγωγής ε, μπανάνας ανέβαζαν ή κατέβαζαν κυβερνήσεις, κατοδοκούν όταν κυβερνήσεις τους ενοχλούσαν ε, γιατί προσπαθούσαν να τηρήσουν τα ελάχιστα εργατικά δικαιώματα ή να ανεβάσουν τους ελάχιστους μισθούς, χρησιμοποιούσαν ακόμα και πραξικοπήματα. Σε αυτές τις χώρες συνεχίζεται η παραγωγή μπανάνας από τις ίδιες εταιρείε ε, και η καταστροφή των δασών, του περιβάλλοντος, ε, άθλιες συνθήκες εργασίας, αλλά και χρήση φυτοφαρμάκων που είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καθημερινές πρακτικές. Την ίδια στιγμή, ε, λόγω αυτών των πολυεθνικών, καταναλώνουμε κατά 99% ένα είδος ε, μπανάνας, όταν υπάρχουν ε, μερικές χιλιάδες είδη μπανάνας. Και αυτό το είδος, ακριβώς λόγω της μονακαλλιέργειας, αυτή τη στιγμή απειλείται με συγκεκριμένη ασθένεια τα μέτρα υποστήριξη των χωρών τη αφρική καραϊβική και του ειρηνικού ήταν πάρα πολύ σημαντικά και η μείωσή του ε, θα αλλάξει πάρα πολύ την πραγματικότητα για του παραγωγού των χωρών αυτών χώρε πολύ φτωχέ που χρειάζονται τη βοήθειά μα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη αγορά μπανάνας παγκοσμίω και η πιο επικερδής. Στα επόμενα χρόνια θα δούμε πραγματικά αυτές τις τεράστιες πολυεθνικές να προσπαθούν να κυριαρχήσουν πλήρω στην αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οθώντα την έξοδο του μικρότερου παραγωγού. Και χρειάζεται πραγματικά την προσοχή μα, η Επιτροπή να είναι σε επιφυλακή για την αυστηρή τήρηση τη ευρωπαϊκή νομοθεσία ανταγωνισμού, κανόνων ανταγωνισμού, ώστε να αποτρέψουμε ε, τι μεγάλε πολυεθνικές να κάνουν κατάχρηση τη δεσπόζουσα θέση του στην αγορά, κατεβάζοντα τεχνητά τι τιμέ στην αρχή προκειμένου να εξαντλήσουν του μικρού παραγωγού και με δημιουργία καρτέλ στη συνέχεια να ανεβάσουν κοστίζοντας πολύ ακριβά ε, για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Αρσένη. Εκ μέρους της ομάδας των Πρασίνων Ελεύθερης Ευρωπαϊκής Συμμαχίας η κυρία Γκρέζα. Σε ό,τι αφορά την έγκριση των εμπορικών συμφωνιών στον τομέα της Πανανά, η ομάδα των Πρασίνων ε, θα τοποθετηθεί κατά. Αυτές ε, οι συμφωνίες ε, ενισχύουν τη δεσπόζουσα θέση των μεγάλων αμερικανικών πολυεθνικών ε, που ήδη ελέγχουν πάνω από 80% της παγκοσμίας αγοράς. Η έγκριση τέτοιων συμφωνιών σημαίνει ότι πηγαίνουμε κατά των χωρών και, των πλέον απομακρυσμένων περιοχών και πάλι θα είναι μικρή παραγωγή που θα νιώσουν τον αντίκτυπο. Οι κανόνε του Διεθνού εμπορίου θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να εγγυθούμε την ανάπτυξη μία τοπική παραγωγή για όλου και την επιστηστική κυριαρχία. Τα χρηματοοικονομικά μέτρα που προτείνει η Επιτροπή για τη Στήριξη των Παραγωγών δεν αρκούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δεσμευτεί όχι μόνο στο να διεξάγει μελέτη αντικτύπων για αυτέ τι συμφωνίε, αλλά και να τροποποιήσει την νομοθεσία τη για να ε, προωθήσει βιώσιμε οικονομίε και τη σχετική παραγωγή. σα. ευχαριστώ. Ευχαριστώ εκ μέρου τη Ομοσπονδιακή ομάδα των... Ε, αριστερά στην Ευρώπη, κύριο Σουαγού. <coughs> Για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, δεν είναι θετικές για μένα αυτές οι συμφωνίε. Αποτελούν την απόδειξη ότι ο μικρός παραγωγός μπανάνας βρίσκεται σε ομοιρία. Είτε πρόκειται για αποκοσμοπισμένε περιοχέ, είτε πρόκειται για χώρε ΑΚΕ. Ο παραγωγό αυτών των περιοχών είναι σε ομοιρία των συμφωνιών τη Γενέβη και των διαπραγματεύσεων τη ΔΟΧΑ που συνεχίζονται. Και αυτέ οι συμφωνίε είναι συμφωνίε που θέλησαν και επέβαλαν και επέβαλε ο Παγκόσμιο Οργανισμό εμπορίων. Η μοίρα των μικρών παραγωγών των ΑΚΕ και των άκρως αποκριμένων περιοχών όντως έχει μικρό ειδικό βάρος έναντι των ισχυρότατων ε, συμφερόντων και των γιγάντων της παραγωγής Αμερικανική Αμερικανικής Υπήρου αλλά και των αντίστοιχων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Και στην αγορά της φάρμας λοιπόν, όπως και στην αγορά της ζάχαρης, εδώ έχουμε την έκφραση μιας ίδιας, μιας ταυτόσιμης κίνησης, μιας κίνησης προς την ίδια παγκόσμια αγορά, η οποία προχωρεί αμήλικτα και συμπιέζει, συνθλίβει τους πιο αδυναμούς και τους πιο μικρούς, τους πιο ευάλωτους. Τέτοιου είδους μέτρα λοιπόν ρύθμιση αγοράς δεν θα μπορέσουν δυστυχώς, Πρόεδρε, να αποτρέψουν τον κίνδυνο της εξάλληψης του μικρού παραγωγού ούτε θα μπορέσουν να σπρώξουν τις χώρες αυτές ΑΚΕ που είναι μεταξύ των πιο φτωχών κρατών του κόσμου προς την ανάπτυξη και την πρόοδο. Θα ήταν σκόπιμο εάν ε, είχαν τη βούληση να διασώσουν και το περιβάλλον και τα εργασιακά δικαιώματα και το βιωτικό επίπεδο των λαών όλοι αυτοί οι ταγοί που σπρώχνουν για την υπογραφή των συμφωνιών της Γενέβης και τότε νομίζω ότι ο κόσμος θα ήταν πολύ πιο βιώσιμος από ό,τι τώρα. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους της ε, ομάδας Ευρώπης των Ελευθεριών και των Δημοκρατιών ο κ. Κάμπιλ Μπάνερμαν για ένα λεπτό. Πρόεδρε, η μπανάνα αυτή αποτελεί το τη ράβδο του πολέμου που μένεται μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης εδώ και 60 χρόνια και τώρα τη χάσαμε παταγωδός στη μάχη, αυτόν τον πόλεμο αυτό τον χάσαμε παταγωδός. Πέσαμε θύματα του, Ευρωπαϊκού, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και υποχρεούμεθα να κατεβάσουμε τα χέρια και να μειώσουμε τους δασμούς μας. Δηλαδή, προσπαθώντα να διασώσουμε τι γαλλικέ απικίε, και μάλιστα εδώ σα δείχνω μια μπανάνα την οποία αγόρασα εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο σούπερ μάρκετ, ε, η οποία όμω δεν ακολουθεί τι ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ ω προ το σχήμα, το μήκο, το φάρδο και την καμπύλη τη ε, Ευρωπαϊκή Μπανάνα. Τέτοιες ανόητε διατάξει ήταν αυτέ οι οποίε έχουν ε, επιβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποδεικνύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι για δέσιμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η πρόεδρο. κυρία Στάσεν τώρα για ένα λεπτό από τους μη Κυρία Πρόεδρε, για δεκαετία η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθούσε μια προστατευτική πολιτική και στον τομέα της μπανανάς. Προστατευτική εμπορική πολιτική ιδέα είναι να διατηρηθούν οι αμερικανικέ εταιρείε εκτό και να βοηθηθούν άλλε χώρε, λιγότερο ανταγωνιστικέ. Όμω ε, τα περισσότερα χρήματα πηγαίνουν στι πλέον απομακρυσμένε περιοχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και Πάρα πολλές φορές ε, ε, κατηγορήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση στον ΠΟΕ γι' αυτό. Πάντοτε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να υποχωρήσει έναντι σε άλλους. Ε, όταν όμως πρόκειται για θέματα ευρωπαϊκά, ουσιαστικά κάνουμε ότι δεν βλέπουμε ο Ευρωπαίος φορολογούμενος πληρώνει για αυτές τις δαπάνες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο. Έτσι λοιπόν καλό είναι να σταματήσουμε με αυτή την πολιτική και να σταματήσει να επιδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές τις οικονομικές αναποτελεσματικότητες. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχουμε τους υπόλοιπους ομιλητές. Ο κύριος Ματάντροβερ για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Κάμπελ, Σίγουρα δεν έρχεται από τα Κανάρια αυτή η μπανάνα που μας δείξατε. Εγώ τώρα θα μιλήσω για την μπανάνα και νομίζω είναι καλό που συζητάμε εδώ για τις μπανάνες και είναι καλό γιατί είναι σημαντικό να επαναλαμβάνουμε ότι πρέπει να προστατεύουμε τους κοινοτικούς παραγωγούς και αυτών, αυτών των Καναρίων. Η σύναψη της Συμφωνίας της Γενέβης δεν είναι καλή είδηση για τους κοινοτικούς παραγωγούς και το ψήφισμα που συζητούμε σήμερα έχει πτυχές Υπότιτλοι AUTHORWAVE που ε, δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικέ σε ό,τι αφορά την προστασία των παραγωγών και από γεωργική σκοπιά. Η Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου έχει διαφορετικά κριτήρια από αυτά που μπορεί να έχω εγώ σε ορισμένε πτυχέ. Γι' αυτό εγώ αξιολογώ τα θετικά και όχι τα αρνητικά. Και είναι θετικό το ότι τελικά τίθεται τέλο τόσα ε, έτη διενέξεων ε, στον ΠΟΕ και επανέρχεται ηρεμία σε ένα τομέα που χρειάζεται σταθερότητα και βεβαιότητα για το μέλλον. Η κοινοτική παραγωγή βρίσκονται σε πλέον απομακρυσμένες περιοχές που έχουν τεράστιες δυσκολίες για την παραγωγή μπανάνας, εξαιρετικής ποιότητας φυσικά, που δεν έχουν καμία σχέση με την παραγωγή μπανάνας άλλων τρίτων χωρών, ε, ούτε σε ό,τι αφορά το κόστος, ούτε το εργατικό δυναμικό, ούτε το σεβασμό του περιβάλλοντος, ούτε ε, των φυτογενομικών εγγύσεων από γεωργική σκοπιά είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η συμφωνία ζημιώνει τους ευρωπαίους παραγωγούς, ε, μειώνεται σημαντικά η δεσμή από τα 176 ε, θα περάσουμε στα 114 και στα 75 για το Περού και την Κολομβία στις σχετικές συμφωνίες. Έτσι λοιπόν μπορώ να σας πω ότι δεν πιστεύω ε, ότι είναι λογικό ότι το 2006 στο ΠΟΣΕΙ προβλέπω όταν ήδη η μείωση αυτού των δασμών. Ε, προβλεπόταν ε, σύμφωνα με τη Συμφωνία της Γενέβης, αλλά ε, ποτέ το 2006 δεν μπορούσε να προβλεφθεί ότι η μείωση του δασμού θα φτάσει μέχρι τα 75 ευρώ όπως προβλέπεται τώρα με αυτές τις συμφωνίες. Έτσι λοιπόν πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες αξιολογήσεις και να θα δούμε ότι χρειάζεται οπωσδήποτε επικυροποίηση του κονδυλίου γιατί ο δασμός των 176 ευρώ θάνατον ο ήδη ήταν ε, χαμηλός. Ε, έτσι λοιπόν οι κοινοτικοί παραγωγοί δεν θα ζητούν τίποτα που να μην είναι αιτιολογημένο και εμεί ως κοινοβούλιο έχουμε την υποχρέωση να του προστατεύσουμε. Το ίδιο και η Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας παρακαλώ. Θα θέλατε να, να βάλετε τα ακουστικά σας παρακαλώ. Βάλτε τα ακουστικά σας. Ευχαριστώ. Μου ζητήσατε το λόγο με την μπλε κάρτα είναι για να λάβετε το λόγο τώρα ή για το καθιστή ε, παρακαλώ να λάβετε υπόψη όμως ότι η μπλε κάρτα είναι μόνο για να υποβάλλετε ερώτηση προς τον υποψήφιο, προς τον ομιλητή. Άρα θα περιμένετε την περίοδο που θα δώσουμε για το καυστιάι. Τώρα η κυρία Στάιλερ παρακαλώ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, να πούμε τώρα για τις μπανάνες του δίκαιου ηθικού εμπορίου, γιατί προέρχονται από από αυτό ευρωπαϊκές φτωχές χώρες και έχουμε εκατομμύρια εδώ τα οποία θα σε Αφρική, σε Καραβική που είναι εξαγωγές χώρες και όλοι αυτοί που δουλεύουν εκεί πέρα ουσιαστικά είναι αντικείμενα εκμετάλλευση από τις πολυεθνικές. Ε, Επομένω, ο κόσμο έχει μπουχτίσει από αυτή τη μεταχείριση και γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σωστό να υπάρχει έτσι ηθικό διοντολογικό εμπόριο, μια που Ξέρετε, για τη Σκοτία είναι το, το πρώτο φρούτο στην κατανάλωση το πιο αγαπημένο και οι ψηφοφόροι μου επίσης ενδιαφέρονται για να είναι ποιοτικό αυτό το προϊόν. Οπότε παρακαλώ συνάδελφοι, μόνο τέτοιες μπανάνες να αγοράζετε. Και να διαδίδουμε στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν κάποια σημεία προστριβής, αλλά θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ευνοήσουμε τους πιο ευάλωτους αυτού του κόσμου ασχολείται με το εμπόριο αυτό. Ευχαριστώ κύριο Σλαβία, είναι ο επόμενο ομιλητή για 1,5 λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, οι διημερεί εμπορικέ συμφωνίε συνήθω είναι ει βάρο των Ευρωπαίων παραγωγών που ε, υφίστανται τι αρνητικέ συνέπειε τη απελευθέρωση. Ε, προβλέπεται τώρα με τι συμφωνίε σε μείωση των δασμών ε, για τι μπανάνε που έρχονται από τι χώρε Λατινική Αμερική. Αυτέ οι συμφωνίε ε, μπορεί να οδήγησαν στο να επιληθεί μια διένεξη δέκα ετιών, όμω θέτουν σε κίνδυνο του Ευρωπαίου παραγωγού και οι συμφωνίε που διαπραγματεύομαστε με τη Λατινική Αμερική σε, ε, μαζί με συνοδευτικά μέτρα για τον τομέα των μπανανών μπορεί ε, να υπονομεύσουν σοβαρά την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαίων παραγωγών. Η υποστήριξη των δικών μας παραγωγών ε, είχε ε, ήταν αντικείμενο εγγύηση μέσω του ΠΟΣΕΙ. Όμω η ίδια μεταρρύθμιση του από το 2006 δεν λαμβάνει υπόψη τη ε, σύναψη αυτών των τελευταίων συμφωνιών. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι είναι κατάλληλο να καλέσουμε το Συμβούλιο ε, να τοποθετηθεί επί τη αναγκαιότητα να έχει χρηματοδοτικού μηχανισμού για να καλύψει τι ανάγκε των Ευρωπαίων παραγωγών, βελτιώνοντα την κατάστασή του και προσπαθώντα να αντισταθμίσει τι ενδεχόμενε ζημίε που θα προέλθουν από την μείωση των δασμών και τη σύνεψη των συμφωνιών. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να ε, προβούμε στην ε, ετήσια αναζήτηση κονδυλίων για να καλύψουμε <coughs> τι ανάγκε των Ευρωπαίων παραγών μπανάνα, αλλά πρέπει να βρούμε μία βιώσιμη λύση που να διαρκεί στον χρόνο για να αποζημιώσουμε του παραγωγού από τι ζημίε του ανοίγματο των αγορών. πολύ, Ύστερα από μια μακρά διελκυστίνδα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης αφετνός και τους Λατινοαμερικανούς παραγούς μπανάνας αφετέρου ε, προχώρησε σε ένα σημαντικό βήμα ε, με τη συμφωνία για τις μπανάνας. Στο πλαίσιο των ε, όρων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Πλην όμω αυτή η συμφωνία δεν, μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Λατινοαμερικανικών κρατών δεν μπορεί να παραγνωρίσει και την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί μπανάνα στις χώρες ΑΚΕ. Είναι πολύ σημαντικό εδώ να, γίνουν, να ληφθούν υπόψη οι εκτιμήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Μπορεί να είναι στοιχειώδης αυτή η απέτηση, αλλά δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε να χαθεί μέρος της παραγωγής από τις χώρες ΑΚΕ ή κονδύλια τα οποία στόχο έχουν να στηρίξουν αυτούς τους παραγωγούς να φτάσουν σε άλλα χέρια. Είτε πρόκειται για αναπτυξιακό ταμείο, είτε πρόκειται για γεωργικά ταμεία. Όλα αυτά τα πράγματα είναι υποσυζήτηση αυτή τη στιγμή και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να εκπληρώσει το καθήκον της έναντι των κρατών ΑΚΕ για να τα βοηθήσει στην ανάπτυξη και το βιώσιμο εμπόριο. Αυτή η συμφωνία λοιπόν έχει παγκόσμια από τα παγκόσμιο αντίκτυπο και ως εκ τούτου θα πρέπει να ρίξουμε και να τη δούμε μέσα από την προοπτική των διαπραγματεύσεων της Ντόχα και θα πρέπει να περιμένουμε αν μετά το 2012 θα αποδειχθεί ότι τα λόγια που ακούμε μετατρέπονται και σε έργα και αν θα μπορέσει αυτή η συμφωνία να αλλάξει κάτι στις συμφωνίες Δόχα. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Σκέλη για ένα λεπτό. Uh, Πρόεδρε, ευχαριστώ. πολύ. Πριν από μερικές εβδομάδες τρελαινόμασταν για τις μέλισσες και τώρα βουίζουμε σαν τις μέλισσες γύρω από την μπανάνα. Το λογοπαίγνω στα αγγλικά με την μπανάνα και τη μέλισσα. Έχουμε όμως ζητήματα και με το περιβάλλον, έχουμε ζητήματα και με τις επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας στον παραγωγό και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να ληφθεί υπόψη γιατί η κύρια ευθύνη η ουδήποτε, η ασδήποτε χώρας, η ουδήποτε φορέα ή οργανισμού είναι να προστατεύσει πρώτα αρχικά το δικό του παραγωγό και μετά να απλώσει χείρα στους λοιπούς. Το ίδιο ισχύει και για την παραγωγή του βόρειου κρέατος. Πολλοί είναι αυτοί που φοβούνται ότι τέτοιου είδους συμφωνίες μπορούν να αποδιοργανώσουν τον τομέα του βοήου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, ναι, αλλά μόνο εφόσον πρώτα προστατεύουμε τους δικούς μας παραγωγούς. Ευχαριστώ πολύ. Κάτσε τη ΆΕ τώρα, κύριε Στατζέρα. Ένα λεπτό όπως πάντα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Βουλευτέ, ήδη με έχετε ακούσει να τοποθετούμε σε αυτό τον οίκο και θα ξαναπώ οι πλέον από απομακρυσμένε περιοχέ από όπου το προέρχομαι δεν έχουν ε, καμία αντίρρηση ούτε τη σύναψη των συμφωνιών τη Γενέβη ούτε των, ε, ούτε των άλλων συμφωνιών που συνήφθησαν εκ των υστέρων. Ε, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι αναπόφευκτε αλλά και σημαντικέ. Όμω πρέπει να πούμε ότι και σε αυτέ τι συμφωνίε υπάρχουν νικητέ και τιμένοι και σε αυτέ τι συμφωνίε συγκεκριμένα οι πλέον μικρισμένες περιοχέ είναι οι τιμένοι και ζημιώνονται. Δεν μπορώ να όπως έκανε και η Κομισιόν σήμερα, επιμένουμε ε, στο επιχείρημα ότι η αναθεώρηση του ΠΟΖΕΙ το 2006 ήδη προέβλεπε αυτή την ε, κατάσταση και ήδη είχαν αντιποζημιωθεί οι παραγωγοί ενώ γνωρίζουμε ότι το 2006 ε, μιλούσαμε για 176 ευρώ τότε ενώ μιλάμε για 114 ε, ευρώ ή ακόμη και 75. Εδώ μιλάμε ε, επομένως για μέτρα αντιστάθμισης. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Έχουμε ένα λεπτό για το Catch Ο κύριος ε, Φερέιρα τώρα έχει δυνατότητα να μιλήσει. Ε, ήθελα να πω ότι αυτοί που θέλουν να κλείσουν στις Αμερικανικές πολυεθνικές ε, τις πόρτες ευρωπαϊκές αγορές που ήδη ελέγχουν το 80% του παγκόσμιου εμπορίου να σε αυτές τις συμφωνίες θα έχουν σημαντικές συνέπειες. Η οι Ευρωπαίοι παραγωγοί, από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ισπανία που το 2008 ήταν υπεύθυνη για την προμήθεια 60.000 τόνων στην ευρωπαϊκή αγορά θα θυγούν οι ίδια η εισηγήτρια δέχεται ότι απειλεί την ύπαρξή τους στο μέλλον η συμφωνία αυτή έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρό που η Κομισιόν ενώ γνωρίζει τις συνέπειες δεν προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα στήριξη στους ευρωπαίους παραγωγούς με ε, αλλαγή του κανονισμού ΠΟΖΕΗ και των κονδυλίων που είχαν εγκριθεί το 2006 μάλιστα και οι χώρες ΣΑΚΕ τις οποίες δεν διαβουλεύτηκαν πριν τη σύναψη των συμφωνιών θα θυγούν σημαντικά ε, και τα παρηγορητικά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί δεν θα ε, αλλάξουν τις συνέπειες αυτές ε, και εδώ δεν έχει καμία, κανένα νόημα να ερχόμαστε και να λέμε ότι ανησυχούμε και να θέτουμε τις ανησυχίες αυτές με τις μορφές, με τη μορφή ανησυχίας. Η Πρόεδρος, αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ θα επισημάνω ε, ότι αυτές οι ομιλίες catch the eye διαρκούν ένα λεπτό αλλά δεν μπορούν να αποτελέσουν μια πλήρη ομιλία και συγχαίρω τη γερμανική καμπίνα για την εξαίρετη απόδοσή της. Παρακαλώ όμως να μην προσπαθείτε αγαπητοί συνάδελφοι εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι σας δίνω το χρόνο να προσπαθήσετε να βάλετε μια ομιλία μέσα σε ένα λεπτό και μόνο. Το λόγο έχει τώρα ο Επίτροπος κύριος Τσόλος. Εσείς έχετε το χρόνο σας και παρακαλώ στο δυνατόν πιο κατανοητά να μας δώσετε την ομιλία σας. Ναι κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω όσο πια μου γίνεται να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις. Γιατί μιλήσαμε για το πώς θα επιληθεί αυτή η διαφορά ή στα πλαίσια των πολυμερών συμφωνιών για δε, τις διμερείς συμφωνίες, δηλαδή με τις χώρες Κεντρικής Αμερικής και Λατινικής Αμερικής εκεί πρόκειται για άλλη ιστορία διότι και σε αυτή την περίπτωση και εκεί έχει συμφέρον να έχει επιθετική ενεργητική δυναμική στάση η Ευρωπαϊκή Ένωση και επίση στη συνέχεια υπήρξε η άλλη παρατήρηση που αφορούσε τις πολυεθνικές ε, οι οποίες κερδίζουν στις χώρες εκείνες και δεν γίνεται αυτό με τρόπο δίκαιο τσακεύμα. Δεν είναι δυνατόν εμεί όμω να γίνουμε κυβέρνηση, γιατί πάρα πολλά θα μπορούσαν να γίνουν εάν τα χρήματα τα οποία δίνονται τελικά απορροφούνται με σωστό τρόπο, αξιοποιούνται με σωστό τρόπο. Επίση αυτό αφορά και τις ε, χώρε που παράγουν ε, μπανάνα και τι απότερες περιφέρειες, τι απομακρυσμένε περιοχέ ε, να σα δείξω τα στοιχεία, κύριε, που το ρωτήσατε αυτό, διότι το 2006 πέραν αυτού του πακέτου που είχε προβλεφθεί κάναμε κάποιο είδου υπολογισμού. Να, έχω εδώ τα στοιχεία. Είχαμε προβλέψει πτώση τη τάση 176 με 137 ευρώ ή το 2009 και επίση τότε θεσπίσαμε την δυνατότητα κατά τι διαπραγματεύσεις της Ντόχα που δεν ξέραμε ακόμα τα αποτελέσματα να είναι δυνατόν ο σχετικός τόρος να πέσει μέχρι τα 79 ευρώ ανά τόνο και γι' αυτό Έχουμε 246 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το πακέτο ΠΟΣΕΙ και 8,4 προσθέσαμε, δηλαδή 22 εκατομμύρια ευρώ ετησίως επιπλέον τόσο ώστε να μπορούμε να προλάβουμε τις ενδεχόμενες επιπτώσεις και για αυτό και ο προπολογισμό του ΠΟΣΕΙ το 2006 ήταν πολύ παραπάνω σύμφωνα με τις επιπτώσεις σε σχέση με την πραγματική συγκυρία του 2006 δηλαδή είπαμε Οπότε πάει αυτό. Να δούμε τι θα γίνει τώρα για άλλου είδου. Ε, αντιστάθμιση και έχουμε μέσα τον σχετικό κανονισμό για το ποσί το οποίο τώρα τον συμφωνούμε με το Συμβούλιο και ίσως θα υπάρξει αντιστάθμιση αλλά ένα μεγάλο κομμάτι που ήδη έχει εκταμιευθεί και σα το είπα ότι υπάρχουν υπολογισμοί και στοιχεία και έχουν γίνει επαφές με τα μέλη. οπότε τα λέμε όλα αυτά τεκμηρωμένα και τώρα όσον αφορά τους μικρούς παραγωγούς. Για τους τις περιοχές έχουμε τους παραγωγούς που θα πρέπει να τύχουν προστασίας. Τι θα γίνει με τους πόρους του ΠΟΣΕΙ, θα πρέπει για αυτούς να διατεθούν. Δεν ισχύει αυτό πάντα και επομένως κάποια στιγμή για το ΠΟΣΕΙ θα πρέπει να γίνει μια προσαρμογή ούτως ώστε ισχυρικοί πόροι πραγματικά να βοηθούν εις αναδιάρθρωση του κλάδου αλλά τα χρήματα τα οποία ήδη έχουν δεσμευτεί για το ΠΟΣΕΗ σαν αντιστάθμιση αν θέλουμε να πάνε σαν ενίσχυση στην αναδιάρθρωση ε, ίσως σε κάποια χρόνια να υπάρξει κάποια εναλλακτική λύση στους μικροπαραγωγούς γιατί θα πρέπει να μην ξεχνάτε ότι εγώ είμαι ανοιχτό σε νέες λύσεις και ιδίως όσον αφορά το ΠΟΣΕΗ ούτως ώστε να χρησιμοποιηθούν καλύτερα αυτοί οι πόροι και Επίσης, θέλω να απαντήσω στον κύριο Κάμπελ που διαφωνεί όσον αφορά την αντιστάθμιση γιατί εκεί στις απότερες περιφέρειες και αυτοί είναι Ευρωπαίοι και αυτοί είναι φορολογούμενοι και μου φαίνεται φυσιολογικό να υποστηρίζονται εάν είναι για λόγο θεμητό. Ναι, αλλά αν γινόταν αυτά που λέτε εσεί, δεν μπορούσατε να αγοράσετε την μπανάνα. Γι' αυτό τα κάνουμε αυτά που κάνουμε. Και γι' αυτό και υπάρχουν ίσως συγκεκριμένου κανόνε οι ευρωπαϊκέ μπανάνε αυτά θέλω να σα πω. Νομίζω ότι χτενήσαμε τα βασικά σημεία. επίση ε, υποτύπων συμπεράσματα πρέπει να σας πω ότι ε, με τι συνομιλίε για το πώς ε, είμαι ανοιχτό να διαπιστωθεί με, τα συγκεκριμένα στοιχεία τη τραπέζη, με ποιο τρόπο οι υπάρχουσες αντισταθμίσεις ή άλλες τυχόν θα μπορούσαν να καλύψουν αυτές τις ανησυχίες όμως θα πρέπει να σας πω ότι πρόκειται για μια συμφωνία που όπως μας ανέφερε η συγγήτρια είναι λέγω συμφωνία που μας βοηθά από πολλές πλευρές και έτσι επιλύεται, διεκπεριώνεται μια προστριβή, μια διαφορά παλιά. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία για το συμβούλιο σας παρακαλώ να το λόγο. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου, ιδιαίτερο ότι όμω ότι πολλέ από τι από τις απορίες, αντιρρήσεις και επιφυλάξει που είχαν εκφραστεί με τι παρατηρήσει των ε, κυρίων και κυρίων βουλευτών ε, απαντήθηκαν. Και θα ήθελα να δώσω και εγώ πλευρά μου κάποιες θέσει. Ε, αν αναλογιστούμε τι είδου ενισχύσει προβλέπεται να χορηγηθούν για να αντισταθμιστούν οι διατάξει και τα μέτρα που εισάγονται προς τα, τα στον τομέα της μπανάνας. Για να στηριχθεί λοιπόν ο παραγωγός από, το, από τις συνέπειες της κατάργησης του, συστήμα, καθεστώτος που ίσχυε μέχρι τώρα νομίζω ότι είναι πολύ ικανοποιητικά αυτά τα μέτρα. Επίσης ένα δεύτερο ζήτημα είναι τι θα συμβεί ε, όταν συνεχιστεί η απελευθέρωση τομέα και καταργηθούν ή μειωθούν ακόμη περισσότερο οι δασμοί. Εν προκειμένου, θα ήθελα να σας ε, αναφέρω ότι το Συμβούλιο σκοπεύει ε, να ξανασυζητήσει το κατά πόσον θα πρέπει να διατηρήσει την υποστήριξή του προς ε, τις χώρες των Άνδρων και της Λατινικής Αμερικής για τέτοιου είδους συμφωνίες στον βαθμό που θα υποβάλει και τις σχετικές προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η σύναψη συμφωνία στον τομέα της μπανάνας αποτελεί το κατακληκτικό βήμα ενός προβλήματος που μας έχει ταρανίσει 15 χρόνια. Και πιστεύω ότι στέφεται με επιτυχία και στις επιτροπές, στι διεθνεί διαπραγματεύσει και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του κύκλο τη Δόχα, βλέπω ότι πρέπει να δοθούν απαντήσει σε όλε τι ανησυχίε που ακούστηκαν σήμερα εδώ και ιδιαίτερα με μέλημα τις ανησυχίες και τους φόβους των πιο ευάλωτων κρατών που πάντα έχουμε υπόψη. Πάντως, οτιδήποτε δεν άπτεται άμεσα το δικού μου πεδίου δεν μπορώ να το δείξω, αλλά νομίζω ότι είναι πλήρη η που παρέχεται με το καθεστώ αυτό και καλό το Κοινοβούλιο αύριο να εγκρίνει το νέο καθεστώ στον τομέα τη μπανάνα. Η πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε τώρα και πάλι την εισηγήτρια. Και συντάκτηρα προφορική ερώτηση, κυρία Παντζάνη, για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και εν μέρη έθεσε και πάλι νέους φόβους και, και πάλι φόβους και ερωτήσεις που είχαμε ήδη συζητήσει στην Επιτροπή. Θέλω να υπογραμμίσω κάτι σημαντικό που νομίζω ότι πολλές φορές ξεχνάμε αυτές τις συμφωνίες ε, αποτελούν ε, την θέση εφαρμογή μια συγκεκριμένη δέσμευση ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι μέλο του ΠΟΕΣ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Πρόκειται για συμφωνίες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει να επιλύσει ένα σοβαρό πρόβλημα με πολλές χώρες, ε, με σημαντικές χώρες και ε, βρέθηκε στο ε, προβληματική αυτή κατάσταση γιατί είχε παραβιάσει την αρχή της μη εισαγωγή διακρίσεων. Έτσι λοιπόν πρέπει να συμβούμαστε τις υποχρεώσεις μας ως μέλος του ΠΟΕ. Και μία συμφωνία εντάσσεται στην επίλυση διαφορών ε, και ε, σε ένα κλίμα το οποίο ζημιώνει και άλλους και πρόκειται μια μία οριστική συμφωνία η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει νέα ισορροπία και το πράττει το είπαμε και το έχουμε γράψει και στην έκθεση με ιδιαίτερη προσοχή έναντι χωρών που βρίσκονται σε λεπτή θέση ως προς την ανάπτυξη. Τα συνοδευτικά μέτρα σίγουρα θα είναι αντικείμενο εποπτείας και θα έλεγα ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό ζήτημα. Το να έχουν προβλεφθεί συνοδευτικά μέτρα είναι σημαντικό, αλλά θα είναι και πιο σημαντικό να έχουμε και τις αξιολογήσεις αντικτύπου για τη λειτουργία τους, να έχουμε τη δέσμευση και είμαι ικανοποιημένη γι' αυτό, τη δέσμευση που ακούσαμε να λαμβάνουν σήμερα και η Κομισιόν και το Συμβούλιο να μην ε, ε, χάσουμε ποτέ την δυνατότητα παρέμβασης με διαφορετικά μέτρα αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Το ίδιο το ΠΟΖΕΙ έχει συμπεριληφθεί στο ψήφισμα ως ένα λεπτό σημείο γιατί και αυτό ε, πρέπει να είναι υποέλεγχο, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η νέα κατάσταση των πλέον απομακρυσμένων περιοχών. Έτσι λοιπόν και αυτό ο αντίκτυπος των συμφωνιών στι ευρωπαϊκέ πλέον απομακρυσμένε περιοχέ που παράγουν μπανάνε, θα είναι αντικείμενο παρακολούθηση και προσοχή. Το Συμβούλιο πλέον αναφέρθηκε στο εξή και είμαι ικανοποιημένη γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα. Την αναγκαιότητα να εργαστούμε ε, για τη διαφάνεια της ε, αλυσίδα εφοδιασμού, γιατί εδώ μιλάμε για την παραγωγή αλλά και για τη διανομή των μπανανών στο εσωτερικό της Ένωσης. Έτσι λοιπόν πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν στο μέλλον, παρακολούθηση της ισχύω των συμφωνιών, της λειτουργίας των συνοδευτικών μέτρων, της καταλληλότητας του ΠΟΖΕ για την προστασία των ευρωπαίων παραγωγών και να χρησιμοποιήσουμε και άλλα μέτρα όπως της διαφάνειας της αλυσίδας εφοδιασμού και να ε, καλύψουμε και την ε, αλυσίδα της διανομής γιατί τελικά έχει συνέπεια στην τιμή των τροφίμων και στην προστασία των καταναλωτών. Αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη όπως και πολλά άλλα συμφέροντα που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση όμως ε, ε, σε όλα αυτά όπως και η προστασία των καταναλωτών θα πρέπει να ξεκινούν από ένα προσδιορισμό της σημερινής κατάστασης από ένα προσδιορισμό της ολοκλήρωσης αυτών των διαφορών. Η Ευρώπη ε, ε, συνάπτει συμφωνία με ε, τις Ηνωμένε Πολιτείες και τις χώρες της Ελληνικής Αμερικής. Έτσι λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να εγκρίνθουν αυτές οι συμφωνίες έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα εργαλεία της αγοράς των μπανάνων και πρέπει να διασφαλίσουμε και τα συμφέροντα των καταναλωτών που έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια της αλυσίδας εφοδιασμού και αν ε, δεν έχουμε ένα σταθερό σημείο αφετηρίας της επίλυσης των διαφορών στον ΠΟΕ όπου ανήκει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να γίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σε ολοκλήρωση της συζήτησης έχουμε πρόταση ψηφίσματος, η οποία θα ψηφιστεί αύριο το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ και τώρα έχουμε μια